διάταξη που είναι προφορικές ερωτήσεις. Αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πέντε συντάκτες έχουμε των ερωτήσεων και θα πάμε με τη σειρά. Πρώτος ο κύριος Σταγιάννη για δύο λεπτά παρακαλώ. Yes. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Κύριε Επίτροπε, αυτή η ερώτηση έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη διαδικασία αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων που είναι ουσιαστικό μέτρο για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση. Η ΜΜΕ είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας ε, και ε, ουσιαστικά κινούν το 55% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος και δίνουν δουλειά σε 80 εκατομμύρια πολίτες. Για να συνεχίσουν όμως να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη θα πρέπει να υποστηριχτούν με χρηματοδοτήσεις που να τους επιτρέπουν ε, να έχουν ένα διεθνή ρόλο, να επενδύουν σε νέα έργα και να προσλάβουν ω υπαλλήλου. Για να πετύχουν αυτό το στόχο δεν αρκεί όμω η νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, μπορούν να υποστηρίξουν πολιτικέ ε, για την πραγματική οικονομία, αλλά δεν μπορούν να τι αντικαταστήσουν ε, για να αντιμετωπίσουν ε, τον πληθωρισμό ε, και ε, την ετελμάτωση της Ευρώπης ε, χρειάζονται μέτρα όπως ο συντελεστής υποστήριξης ουσιαστικά βοηθά το να βρουν την ισορροπία. Χάρη σε αυτό το συντελεστή υποστήριξη το τελευταίο 1,5 χρόνο η τραπεζική επίστοση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε 2% έναντι της μείωσης του 7% σε σχέση με αυτά που δόθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις και μειώθηκαν κατά 20 βασικές μονάδες τα επιτόκια. Εμείς ζητούμε ο συντελεστής υποστήριξης να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί και σε πιστώσεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι λοιπόν να εξαλείψουμε το κατόφλι που υπάρχει σήμερα. Αυτό θα επέτρεπε σε περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως μεσαίες, να επωφεληθούν από το συντελεστή υποστήριξης. Επίσης, Επίσης υποστηρίζω και τη δέσμευση του Επιτρόπου Χιλ να καταστήσει αυτό το μέσο σε ένα διεθνές πρότυπο μέσω της Επιτροπής της Βασιλείας. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φερέιρα, αλλά δεν τη βλέπω. Οπότε θα προχωρήσουμε στην κυρία Λόπες για δύο λεπτά παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η δική μου, όπου τα οικονομικά συμφέροντα έχουν καταφέρει τεράστιο πλήγμα στις χαμηλές κοινωνικές ε, τάξεις με μεταρρυθμίσεις που διέριξαν πλήρως το κοινωνικό ιστό πριν από την κρίση. Και αυτή η διαδικασία εξηγεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σήμερα. Έχουν εξαφανιστεί οι περιφερειακές τράπεζες, έχει συγχωνευτεί ο τραπεζικός τομέα και δεν δίνει καμία τραπεζα γιατί τα κρατάει τα χρήματα για να τα τζογάρει στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, όμως είναι αυτές που ε, παράγουν και δίνουν τοπική απασχόληση και δεν ενδιαφέρουν ε, τα σύγχρονα Golden Boys. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως να ε, πάνε στο χρηματιστήριο για να αποκτήσουν κονδύλιο, κονδύλια και έτσι θα εκτεθούν ακόμα περισσότερα στους κινδύνους των διεθνών χρηματοπιστωτικών. Οι εργαζόμενοι πέφτουν θύματα της ανεργίας, βλέπουν τους μισθούς τους να περικόπτονται. Είναι αβέβαιος ο ορίζοντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ότι όλες οι θέσεις εργασίας γίνονται όλο και πιο αβέβαιες ε, είναι ένα εργαλείο για να επικρατήσουν στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων όμως ε, είναι απαραίτητη για να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγορά για τα προϊόντα τους. Έχουμε τεχνική συζήτηση ενώ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει ήδη πει ότι ελάχιστα θα προκύψουν από αυτή τη συζήτηση. Ας ε, συζητήσουμε ειλικρινά για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την τελμάτωση, για το βάλτο στον οποίο έχετε ρίξει εσείς όλες αυτές τις χώρες με τις πολιτικές σας λιτότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτικές που θα μεταμορφώσουν το οικονομικό τοπίο, θα συνάψουμε συμμαχίες με τον κοινό μας εχθρό που είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ευχαριστώ κύριε πολύ κύριε Πρόεδρε και Στόγιο. Ε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε ε, στην ε, έγκριση της οδηγίας ε, και του κανονισμού του τέταρτου για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, το Κοινοβούλιο σωστά ζήτησαν να μειωθούν οι κεφαλαϊκές απαιτήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε μια έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας που διαπιστώνει ότι σε νέα κράτη-μέλη που ελέγχθηκαν ε, δεν συνάδουν με το πλαίσιο της Βασιλείας ε, οι τράπεζες ε, και αυτό μας έχει ανησυχήσει. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να διατρανώσουμε ότι οι μικρότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι απολύτως απαραίτητο για να μπορούν στο μέλλον να χρηματοδοτούνται. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουν δυσκολίες χρηματοδότησης οι μικρομεσαίες. Έχουν και παρά έχουν, όχι μόνο στην περιφέρεια, ακόμα και στις χώρες που αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά εύρωστε. Υπάρχουν εταιρείες που δυσκολεύονται πάρα πολύ να έχουν πρόσβαση σε δάνεια. Και λόγω του γεγονότος ότι το 99% ε, των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και 23 εκατομμύρια είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν. Στο μέλλον χρειάζεται δανειοδότηση γιατί και με την Ένωση των Κεφαλαίων δεν μπορούν ε, να χρηματοδοτούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις απρόσκοπτα. Ε, οι φιλελεύθεροι και δημοκράτες, η πολιτική μας ομάδα συμφωνεί και καλεί με το υπόλοιπο κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει έναν τρόπο και έναν δρόμο έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη δανειοδότηση εξασφαλισμένη οι μικρομεσαίες. Γκρινιάζουν οι τράπεζες και διαμαρτύρονται για την υπερβολική ρύθμιση. Ε, το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη που λέει ότι και οι μικρομεσαίες τράπεζες ε, εδώ είναι σε μειονεκτική θέση. Παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί και ε, τις θέσεις εργασίας και να μην εγκαταλείψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σουίνμπορν. Thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης και της δικής μου περιφέρειας έχουν δείξει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα, αλλά τώρα χρειάζονται κεφάλαιο για περαιτέρω μεγέθυνση στα πλαίσια του ε, κανονισμού που διαπραγματεύτηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Δόθηκε έμφαση σε υψηλές κεφαλικέ απαιτήσει για τα πιστωτικά ιδρύματα, όμως ε, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό στην πραγματική οικονομία. Ένα μέρο αυτών των μέτρων ήταν τη υποστήριξη των ΜΜΕ για να δοθούν κίνητα στι τράπεζε να δανείσουν στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση της EPA για την εφαρμογή μας δείχνει ότι είναι μικρός ο αντίκτυπος και παραθέτω ο δανεισμός από τις τράπεζες έχει μειωθεί σημαντικά σε όγκους 95 δισεκατομμύρια έπεσε το 2014 ε, όμως ε, η, ανάλυση της CBA της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα όλου του συντελεστή υποστήριξης για τις ΜΜΕ όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να το δούμε αυτό μεμονωμένο καθώς υπάρχουν και άλλοι συντελεστές που πλήττουν την, το δανεισμό όπως ε, και το θέμα της εμπιστοσύνης και μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων. Όμως βάσει δεδομένων που έχουν αναλυθεί από την Τράπεζα της Αγγλίας μας λένε ότι το 97% των ΜΜΕ ε, που ζήτησαν δάνεια τα έλαβαν οι έρευνες της ε, EBA εξετάζουν μόνο το θέμα του εφοδιασμού σε κεφάλαιο και πρέπει αυτό να το δούμε κάπως με σκεπτικισμό η Κομισιόν θα πρέπει να δει τα ευρύτερα θέματα εμπιστοσύνη στον τομέα των ΜΜΕ και να έχει αυτά τα θέματα κατά νου όταν θα αναθεωρήσει το συντελεστή υποστήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα καλούμε τον Επίτροπο Χάν να απαντήσει. Uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πείγνωση τη σημασία του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στην οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτω προσιλωμένη στην κατεύθυνση αυτή για να βρει τι κατάλληλε πολιτικέ και τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε χρηματοδότησή του. Έχουν πρόβλημα και εμπόδια διαρθρωτικά αυτή τη στιγμή, όπω ακούσαμε γιατί εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τη δανειοδότηση των τραπεζών, ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης και πρόσβαση στις κεφαλαίες η εξάρτηση από λιγότερο διαφοροποιημένε πηγέ και από τι τράπεζε καθιστά τι μικρομεσαίες πιο ευάλωτες όταν έχουμε αρνητική οικονομική συγκυρία και ύφεση. Είναι τεράστιε οι δυσκολίε στην Ευρώπη των εταιριών αυτό μετά την κρίση που γνωρίσαμε. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό σε κάποια κράτη-μέλη που οδήγησε σε ανησυχίες και φωνές που ακούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπό το πνεύμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει ε, ε, να συμπεριληφθεί ο συντελεστή υποστήριξη των μικρομεσαίων στι οδηγίε για τι κεφαλαϊκέ ε, απαιτήσει CDR και και για τον κανονισμό επίσης που αφορά τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων. Ο συντελεστής υποστήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 2014 έχει τεθεί σε ισχύ. Χάρη σε εσά και τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναγνωριστεί η σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο του θέματος αυτού και η Επιτροπή Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών τώρα σκέφτεται να ε, μειώσει ε, τις απαιτήσεις για την έκθεση ε, των μικρομεσαίων στην αναθεώρηση του κανονισμού για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει που θα ε, δημοσιευτεί στο τέλη του έτου, θα το λάβουμε υπόψη. Ιδιαίτερα θα δούμε πώς επηρεάζει τον όγκο της δανειοδότησης των μικρομεσαίων ο συντελεστής αυτός από τότε που εισήχθη σε σχέση με άλλους ε, παράγοντες ε, το ιστορικό της δανειοδότησης στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Θα δούμε και θα εξακριβώσουμε κατά πόσο με βάση τα στοιχεία που έχουμε ο συντελεστής υποστήριξης των μικρομεσαίων παραμένει ενισχύει. Θα βαλάβουμε υπόψη πάντα το μέγεθος της εταιρείας και το μέγεθος του δανείου. Έχουμε διάφορες πηγές ε, πληροφόρησης, όπως ήταν και η πρόσφατη δημόσια διαβούλευση των αρμοδίων φορέων. Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε αυτή η διαβούλευση του 2015. Πρόσφατα η ε, Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών, ε, η EBA, ε, δημοσίευσε μια έκθεση και αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τις συστάσεις που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελλοντικά. Στο μέλος... Επίσης, στο μέλλον δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης των μικρομεσαίων τα τραπεζικά δάνεια. Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η χρηματοδότησή τους και οι πηγές τους για να μην κυριαρχούν οι τράπεζες και να μην έχουν τόσο δεσπόζουσα θέση. Αυτό είναι ένας από τους στόχους του σχεδίου Ένωσης των Κεφάλαιων Αγορών για να ενισχυθεί και ο ρόλος τους ε, για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ο κύριος Άλμπου, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, Θέλω να καλωσορίσω τα λόγια του Επιτρόπου. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι κινητήρια ε, δύναμη τη οικονομία και της δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είναι το κέντρο της πολιτικής δραστηριότητας αυτού του οίκου. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για την ε, μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε όχι μόνο τώρα αλλά και όταν ήταν και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υποστηρίξει τις ΜΜΕ γιατί χάρη σε πολλές από τις πρωτοβουλίες ε, που ανέλαβε ο Αντώνιο τώρα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Και όπως είπε ο κύριος Σταγιάννη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι η λύση, αποτελεί μόνο μέρος της λύσης. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι ο συντελεστής υποστήριξης είναι κάτι θετικό, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και προς την ενιαία αγορά κεφαλαίων. Και σας ζητώ, κύριοι βουλευτές, να υποστηρίξετε τα πρώτα νομοθετικά πακέτα που σχετίζονται το θέμα, το πακέτο της τυπλοποίησης και είμαι και εισηγητής. Θα ήθελα να επιταχύνουμε την νομοθετική διαδικασία για να πετύχουμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, την υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ είναι ότι σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χάν για τα λόγια του, καθώς και τον Επίτροπο Χίλ για την απάντηση στην επιστολή που έστειλαν αρκετοί βουλευτέ τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εξέφρασε μία θέση ξεκάθαρη Υπάρχει ευρύτατη πλειοψηφία της Επιτροπής Εκών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι ο συντελεστή υποστήριξη των ε, μικρών και μεσών επιχειρήσεων πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Αυτό είναι ένα πολιτικό δεδομένο και προφανώς η Κομισιόν και τα άλλα όργανα της Ένωσης δεν μπορούν να μην το λάβουν υπόψη ότι εμείς έχουμε μία κάθετη πολιτική βούληση Εμείς ε, διαβάζουμε με πολύ ενδιαφέρον και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όμως ε, αυτό δεν ε, μας αποτρέπει στο να υποστηρίξουμε το θέμα της προληπτικής πολιτικής εναντί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ελήφθη αυτή η πρωτοβουλία και τώρα με σαφήνεια λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντελεστής υποστήριξης. Και θα μπορούσαμε ίσως ε, να αντιστρέψουμε ε, τις αποδείξεις που αναφέρονται εδώ, το χάρη ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με το κίνδυνο για το 1,5% μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να πρέπει να αυξήσουμε και το κατώτατο όριο, όχι να το μειώσουμε. Έτσι λοιπόν ε, εμείς θα συνεχίσουμε την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για το θέμα αυτό και ευχαριστούμε και την Κομισιόν. Ο κύριος Βιέγας, ένα μισή λεπτό. Οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξή τους ε, και την χρηματοδότησή του είναι γεγονός. Πέρα από όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να επιληθούν τα προβλήματα, από το πρόγραμμα COSME, τους ορίζοντες 2000, τον ορίζοντα 2020 μέχρι και ε, τον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων, ε, τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ρηχθεί από την ΕΚΤ στο σύστημα δεν αρκούν. Και ο ίδιος ο ΣΑΤΟ αναγνωρίζει. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πού είναι η ρίζα του προβλήματος. Για μας το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της λιτότητας που υποσκάπτει την εμπιστοσύνη και στο ότι το τραπεζικό σύστημα προβαίνει σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μόνο μια πολιτική δημοσίων επενδύσεων μαζί με μια αναρδιάθρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος θα μπορέσει να οδηγήσει σε ανάπτυξη και να θέσει την οικονομία στην υπηρεσία του ανθρώπου και της ανάπτυξης. Thank you, Mrs. Parker. Ευχαριστώ κυρία Πάρκερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η προφορική ερώτηση αναφέρει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αληθές εν μέρη. Ωστόσο δεν λύνει το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το άχθος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι είναι ε, τεράστιος ο αριθμός των κανόνων τους οποίους πρέπει να ε, πληρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν πιο ψηλές από τη στήλη του Νέλσονα ε, όλες οι νομοθετικές διατάξεις ε, που αφορούν Βρετανούς εργαζομένους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργοδότες. Δεν απορεί κανείς λοιπόν που οι Βρετανικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι σιδηροδέσμιες από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, με την οποία πρέπει να συμμορφούνται και οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις και δεν απορεί κανείς που θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 31 Ιουνίου θα αρχίσει να ανθεί η οικονομία γιατί θα απελευθερωθεί από αυτή την επαχθή γραφειοκρατική νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Ο κύριος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Μικρό. Χωρίς μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Πίπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω για τη Βρετανική οικονομία πραγματικά θα ήταν καλύτερο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ξέρει κάθε επιχειρηματία. Δυστυχώ κάποιοι πολιτικοί δεν το ξέρουν αυτό. Τώρα που έχουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παγκόσμιες εταιρείες και οι παγκόσμιες τράπεζες. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, τότε θα ήταν χαμένοι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς καλά που υπήρχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε διάφορους κλάδους που κατάφεραν να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις ε, ταυτίζονται ε, με την περιοχή τους οι ιδιοκτήτες, με τους εργαζομένους. Μην τους δυσκολεύουμε τη ζωή άχρηστα. Είναι πραγματικά δικαιολογημένο και δίκαιο να υπάρχει συντελεστής υποστήριξης ε, των μικρομεσαίων ε, στην εκτίμηση κινδύνου και στη ε, ίδια κεφάλαια. Είναι πραγματικά εκείνοι που απορροφούν τους κραδασμούς της οικονομίας και των χρηματαγορών. Ο συντελεστής υποστήριξης όχι απλώς θα πρέπει να παγιωθεί, αλλά να αυξηθεί και το όριο και για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει να υπάρχουν και άλλες ελαφρύνσεις όταν πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις και παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη της. Γιατί οι επενδύσεις των μικρομεσαίων επενδύσεις στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Έχετε μπλε κάρτα του κυρίου Ρούμπιχ. Τη δέχεστε. Είναι λίγοι συνάδελφοι. Αλλά βεβαίως ο κύριος Ρούπιχ είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίπερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς πολύ. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βάση για μια καλή χρηματοδότηση είναι τα κέρδη της επιχείρησης. Και αυτό έχει να κάνει και με τη φορολόγηση. Πιστεύετε λοιπόν κύριε Πίπερ ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο που κάνουν τα κράτη-μέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς μικρόφωνο πάλι κύριε κύριος Πίπερ. Φυσικά. Το θέμα της φορολόγησης είναι προφανές. Θα πρέπει να φορολογούνται οι εταιρείες εκεί που παράγουν κέρδη. Γι' αυτό και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή για κάποιες κακές συμπεριφορές και ανάρμοστες των εταιριών και πιστεύω και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα έκανε σε όλα τα νέα θέματα που προτείνει, είτε νέε ρυθμίσεις για το ΦΠΑ, είτε ε, μια κοινή ε, ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των εταιριών, θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί πάντα πάγια ζητάμε και εμείς στο ΕΛΚ ε, μια μελέτη αντικτύπου για τις μικρομεσαίες. Και τώρα στη διαδικασία κάτσε ο κύριος Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ η ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής Το να τι υποστηρίξουμε δεν θα πρέπει να είναι ένα απλό σύνθημα. Η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίε, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ήμουν κι εγώ κάποτε νέο επιχειρηματία. Ποια τράπεζα θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο επιχειρηματία, πώς μπορεί ε, να έχει πρόσβαση επιχείρηση σε κάποιες αγορές ε, αν μόνο οι πολυεθνικές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Αυτό ο συντελεστή υποστηρίξη είναι ένα καλό μέτρο, αλλά δεν επαρκεί. Θα πρέπει και να υποστηρίξουμε και τα startup παραδείγματο χάρη το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Θα επέτρεπε να έχουμε 75 δισεκατομμυρία για τέτοιες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν το 55% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούν εβδομήντα εκατομμύρια πολίτες ενώ για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό δανεισμό. για την ενίσχυση αυτού του δανεισμού από τα πιστωτικά ιδρύματα έχει εισαχθεί στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ως συντελεστής μείωσης κεφαλαίου για τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο οποίος σύμφωνα με ε, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ωστόσο, οι επιπτώσει του συντελεστή στήριξη δεν είναι ακόμα γνωστέ επιπλέον σε χώρες όπως η ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια μόνο το 18% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνει αίτηση για δάνειο ενώ το 38% συναντά αυξημένες δυσκολίες κατά την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. επιπλέον κύριε Χάν στην ελλάδα η τρόικα στην οποία συμμετέχει και η κομισιόν επιβάλλει την πώληση των κόκκινων δανείων non performing loans των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιθετικά funds με αποτέλεσμα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με διάλυση και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Τι λέτε γι' αυτό κύριε Χάν, πώς συμβιβάζονται αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με αυτά τα οποία συζητούμε εδώ. Θα συνεχίσετε αυτή την επιθετική πολιτική ως Τρόικα για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, όσοι είστε ακόμα παρόντες. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη συζήτηση. Λυπάμαι που τέτοιες ώρες συζητούμε τόσο σημαντικά θέματα όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη τόσο αργά. Γιατί πραγματικά είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ήθελα να θυμίσω ότι στην Ευρώπη έχουμε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περίπου άλλους τόσους ανέργους. Και αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάμβανε ένα άνεργο δεν θα είχαμε καθόλου ανεργία στην Ευρώπη. Ας το σκεφτούμε. Και αν, δούμε το αφήσουμε αυτό στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, θα έπρεπε κάθε εταιρεία να προσλάβει καζομένους. Θεωρητικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικές είναι λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται και να ασχολείται εντατικότατα με την εξέλιξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι έχουμε τέτοια προσέγγιση ε, ώστε να δημιουργούμε προϋποθέσεις και να μην έχουμε ε, ε, κάποια χειραγώγηση, να μπορούν να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Εμείς θα τους δίνουμε ένα πλαίσιο, αλλά την πρωτοβουλία, την επιχειρηματική θα πρέπει να τη λαμβάνει κάθε επιχείρηση. Μόνο τότε αναπτύσσεται η οικονομία και έχουμε επιτυχία, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και εξασφαλίζονται και διαφυλάσσονται. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Νομίζω μας δώσατε τροφή για σκέψη. Κύριε Μαριά, σας παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας δεν είναι αναμένο, κύριε Μαριά. Λοιπόν, δεν ξέρω δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει ο Επίτροπος, δεν ξέρω αν επιθυμεί. Αν δεν επιθυμεί, ελπίζω να σέβεστε την απάντησή του. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε. Όχι, καλώς. Σα ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα έλεγα κύριε Επίτροπο, ότι σας δώσατε μας